την έκθεση ΝΟΚ για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. κύριος Χουάν Νόγκ και έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους Σκιώδης και την πρόεδρο της Επιτροπής μου, την κυρία Σάρον Μπόλς, με την οποία συνεργαστήκαμε πολύ στενά. Η έκθεση αφορά την αθώριση του κανονισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα και κύριο στόχο έχει να ενδυναμώσει την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων μέσω της ανεξαρτησίας των στατιστικών υπηρεσιών και της διαφάνειας των διαδικασιών. Δεν σας υπενθυμίζω όλο το ιστορικό. Μία σύνοψη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σοκαριστεί από το μαγείρεμα των ελληνικών στατιστικών στοιχείων και με αφορμή αυτό θελήσαμε να γίνει μια ολόκληρη μεταρρύθμιση βάσει της οποίας η αξιοπιστία των αριθμών θα μας δίνει αξιόπιστα στοιχεία και για μέτρα όπως την εξάμετρο. Six pack. Επομένως, ζητάμε πρώτον ενδυνάμωση του δεοντολογικού κώδικα για περισσότερο αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία στις σχέσεις κομισιών και κρατών μελών. Δεύτερον, να δοθούν εξουσίες και δικαιοδοσίες διευρυμένες για έρευνες από την Κομισιόν. Τρίτον, ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας του Eurostat με διαβούλευση με το Κοινοβούλιο ως προς τον ορισμό του Γενικού του Διευθυντού. Επί αυτών με την προηγούμενη Προεδρία του Συμβουλίου είχαμε συμφωνήσει. Και το κείμενο αυτό αυτή τη στιγμή, αύριο δηλαδή, θα ψηφιστεί. Δυστυχώς η Κομισιόν αντιτίθεται και χρησιμοποιεί τις δικαιοδοσίες που έχει για να το μπλοκάρει, επιβάλλοντας ομοφωνία στο Συμβούλιο. αλλά στο Συμβούλιο υπάρχουν αντιπροσωπείες που θέλουν να ενδυναμωθεί η συμφωνία και άλλες που αντιτίθενται και επομένως δεν πρόκειται να υπάρξει ομοφωνία και είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στο Συμβούλιο σήμερα που η Προεδρία δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε καν και μια καινούργια εντολή για καινούργιο τριμερή διάλογο. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι εθνικές διατάξεις είναι, δεν αρκούν και παρόλα αυτά εμείς ξεπερνάμε την πρόταση και της ε, Κομισιόν για όλα αυτά. Όπως για τους διευθυντές των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Παραδείγματο χάρη, η συμφωνία προβλέπει οι διευθυντές αυτοί να καθορίσουν κατευθυντήριες γραμμές που να εγγυώνται την αξιοπιστία των στοιχείων. Είναι και αυτό μια πρόοδος. Αλλά δεν το λέει η πρόταση της Κομισιόν, η δική μας το λέει. Σε άλλο άρθρο προβλέπεται η ισοτιμή ανδρών και γυναικών στον ορισμό των διευθυντών των στατιστικών υπηρεσιών και αυτό καινούριο. Σήμερα δεν υπάρχει πλειοψηφία για να προχωρήσουμε περαιτέρω στο Συμβούλιο. Μερικά κράτη-μέλη θεωρούν ότι ήδη πήγαμε πολύ μακριά και ο συμβιβασμός αυτός είναι ο καλύτερος δυνατός. Η Κομισιόν αντιτίθεται επίσης στο αίτημα του Κοινοβουλίου για την ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας του Eurostat. Για μας αυτό σημαίνει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο πριν εγκριθεί ο ορισμός του Γενικού του Διευθυντού και να προβλέπονται διαφανείς διαδικασίες πειθαρχικές. Όλα αυτά είναι πρόοδος επί της αρχικής πρότασης της Κομισιόν και δεν θα έπρεπε να αντιτίθεται αυτή. Το Eurostat δεν είναι γενική διεύθυνση της όπως οι άλλες είναι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Γραφείο και αυτό απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ανεξαρτησία. Θα ήθελα να υποβάλω μια ολοκληρωμένη πρόταση για το διμερή διάλογο, αλλά δυστυχώς αυτό είναι αδύνατο για τους λόγους που σας εξήγησα. Γι' αυτό προτείνω αύριο να εγκρίνουμε το κείμενο της πρώτης συμφωνίας με την Προεδρία και να ζητήσουμε έτσι από το Συμβούλιο να τοποθετηθεί πρέπει να προχωρήσει το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και είμαι έτοιμος να ξαναρχίσω τις διαπραγματεύσεις μόλις τελειώσει η ψηφοφορία. Καταλήγω λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα βασίζεται στη συνεργασία και όχι στην επιβολή και επομένως η Κομισιόν πρέπει να πείσει τα κράτη-μέλη για να προχωρήσουμε προς ένα όλο και πιο ανεξάρτητο και διαφανές σύστημα. Αν αποτύχει η διαπραγμάτευση για λόγο της Κομισιόν, αυτό θα αποτελούσε για εκείνη σημαντική πολιτική ήττα. Θα έχανε το ρόλο, τον ηγετικό ρόλο που, έχει, που είχε μέχρι τώρα στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η Κομισιόν θέλει να είναι επικοδομητική και ελπίζω να μπορούμε να της έχουμε εμπιστοσύνη ως εταίρο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Δυστυχώ όμω πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ξεπεράσατε το χρόνο ομιλίας που είχαμε προβλέψει για το τέλος της συζήτησης. Το 1,5 λεπτό που χρησιμοποίησατε δεν θα μπορέσετε να το έχετε στο τέλος. Μόνο 30 δευτερόλεπτα θα σας δώσουμε. Τώρα παρακαλώ τον Επίτροπο Σεμέτα να λάβει το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κύριε Σιγητά. Χαίρομαι για τη σημερινή συζήτηση, διότι όλοι συμμετείχαμε ενεργά σε θαραλές και πολύ σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να έχουμε καλύτερη και βελτιωμένη οικονομική διακυβέρνηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια υπάρχουν νέε προκλήσει που δημιουργούνται για τα επίσημα στατιστικά από αυτέ τι μεταρρυθμίσεις, αλλά οι πολιτικέ μα θα είναι αποτελεσματικέ και αξιόπιστε, εάν έχουμε τα καλύτερα δυνατά ε, στατιστικά στοιχεία, τα οποία να είναι ακριβή και αξιόπιστα. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στα κράτη-μέλη θα είναι αξιόπιστα και θα βασίζονται σε ε, σταθερά ε, και ανεξάρτητα στατιστικά συστήματα και εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Αυτές οι σκέψεις ήταν ε, ο κινητήριος μοχλός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ανέκαθεν τα θεματολόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό κατέστη σαφής και στο σχέδιο έκθεσης το ο οποίο εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα τον περασμένο Δεκέμβριο για το θέμα αυτό. Θα πρέπει βέβαια να ομολογήσω ότι μετά από αρκετές ε, διαπραγματεύσεις ε, η ε, νομοθεσία για τα ευρωπαϊκά στατιστικά έχει χάσει κάποιους από τους βασικούς πιο φιλόδοξους στόχους που είχε αρχικά η πρόταση. Καταρχάς δίνεται έμφαση στην θεσμική δομή, για παράδειγμα τη Eurostat και όχι σε άλλες λύσεις πρέπει να ενισχύσουμε και να διευκρινίσουμε το ρόλο των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών εντός των εθνικών του στατιστικών συστημάτων και να διασφαλίσουμε ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα διατηρήσουν την ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών υπογράφονταν δεσμεύσεις ε, για την ε, ε, αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων. At national Δίνονται στοιχεία ε, στατιστικά σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για όλους όσους συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρηθεί θεσμική ισορροπία, γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα ισορροπίας μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών συστημάτων ως προς τους επικεφαλείς των στατιστικών υπηρεσιών. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δυσκολίες να δεχτεί τις τροπολογίες ε, υπό τη μορφή που παρουσιάζονται τώρα. Κυρίως ε, κάποιες τροπολογίες που αφορούν το Γενικό Διευθυντή της Eurostat. Αλλά είμαστε διατεθειμένοι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ώστε να προσανατολιστούμε προς τη σωστή κατεύθυνση για αυτή τη στρατηγική μεταρρύθμιση και βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας και στο επίπεδο φιλοδοξίας που θα επιδείξετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα η κυρία Γκάλπελτς. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εύχομαι κάθε επιτυχία στον εισηγητή καταρχάς. και ξεκινώ με ένα ουγγρικό ρητικό ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Ποιοι είναι οι καλοί λογαριασμοί λοιπόν. Εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει στατιστικές εσφαλμένες, στατιστικές οι οποίες έχουν οδηγήσει και σε ε, κλειδονισμούς οικονομικούς και κοινωνικούς, θα πρέπει ίσως να δούνε τι σημαίνει ακριβώς καλός λογαριασμός. Γι' αυτό καλό θα είναι να έχουμε ένα σύστημα στατιστικής αξιοπιστής, ένα σύστημα που θα αποτελεί και βάση για τις όποιες πολιτικές αποφάσεις. Η έκθεση αυτή δεν μιλάει μόνο για τη συλλογή στοιχείων, αλλά και για την αξιοποίηση, για, την, ε, για τη θεσμοθέτηση του συστήματος αυτό. Και γι' αυτό και στις στατιστικές υπηρεσίες, τις εθνικές, πρέπει να ε, ληφθεί μέρη ώστε οι διορισμοί να γίνονται ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές επιλογές, πράγμα το οποίο ήδη έχουμε επιτύχει στην Ουγγαρία, όπου διορίζεται για έξι χρόνια παρά ε, ο επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας, ενώ η θητεία του Κοινοβουλίου μας είναι τετραετής. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα σύστημα το οποίο να ξεπερνά ή να εξαντλεί τα όρια του δικαίου και δεν μπορεί να ασκούνται πολιτικές επιρροές στις στατιστικές αυτές. Βεβαίω, μπορούν και οφείλουν να προσφέρουν το συνδρομή τους οι κρατικές αρχές στις στατιστικές υπηρεσίες για τη συλλογή των δεδομένων. Γι' αυτό και θεωρώ απαραίτητο και χρήσιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη της Επιτροπής των Οικονομικών Υποθέσεων να καλέσουν σε ακρόαση τον ε, επικεφαλής της Eurostat. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ποσά μέχρι και 90 εκατομμυρίων ευρώ και πρέπει να είμαστε θέση να τα ε, ελέγξουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Οι επόμενοι δύο μιλητέ δεν βρίσκονται στην αίθουσα αυτή τη στιγμή. Περνάω στη διαδικασία Cars και το λόγο θα λάβει ο κύριο Κέλλη. Παρακαλώ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω στο Προεδρείο κύριε Καρά. Ο κόσμος λέει ότι η στατιστική πάντα ψεύδεται και υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό για άμα χρησιμοποιούνται τα στατιστικά στοιχεία επιλεκτικά. και προσπαθούν ορισμένοι να αποδείξουν τις απόψεις τους με τη στατιστική αντί να προκύπτουν οι απόψεις τους από τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Στον αθλητισμό ιδίω χρησιμοποιείται μεγάλη κατάχρηση, κακή χρήση των στατιστικών στοιχείων για να καλυφθεί η πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε αξιοπιστία και όχι μόνο για τον αθλητισμό αλλά και για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λιπεράτσικη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Διαπιστώνω κάποιες Αντιφάσει μεταξύ της ομιλίας του εισηγητή και των παρατήρησεων της κυρίας Πέλτς γιατί ο εισηγητής παρατηρεί ότι υπάρχουν δισταγμοί βραδιμπορίες ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τον διορισμό στη θέση του επικεφαλής της ε, Στατιστικής Υπηρεσίας. Κυρία Πέλτς, θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, είστε πιο κοντά στις θέσεις του εισηγητή ή του Επιτρόπου, γιατί εγώ προσωπικώς υποστηρίζω τις θέσεις του εισηγητή. Κυρία Τόμασεκ. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι εδώ πρόκειται για ένα θέμα κλειδί. Πρέπει στα στατιστική να είναι αξιόπιστη στα μάτια των πολιτών και να μην γίνεται εργαλείο χειραγώγησης. Ένας Κροάτης υπουργός πρόσφατα ομολόγησε ότι η κυβέρνηση είχε δημοσιεύσει ψεύτικα στατιστικά στοιχεία για να δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξία. Αυτά είναι πολύ άσχημα πράγματα και νομίζω ότι η επιβολή κυρώσεων σε όσους χειραγωγούν τα στατιστικά στοιχεία είναι κάτι θετικό. Μια καλύτερη οργάνωση της στατιστικής, ε, των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών μελών θα ήταν ευκταία γιατί θα μείωνε τις δυνατές χειραγωγήσεις που είναι κάτι τόσο αρνητικό για τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι ερμηνεύω πολύ διασταλτικά τον ε, κανονισμό. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Λιβεράτσκι στη διαδικασία Καρστία, χωρίς να έχει ζητήσει μπλε κάρτα, αλλά διατυπώνοντας ερώτηση στην κυρία Πέλτς, χωρίς προηγουμένως να έχει χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της μπλε κάρτας, παρακαλώ ωστόσο την κυρία Πέλτς να δείξει κατανόηση και μια και αναφέρθηκε προσωπικά το όνομά της να απαντήσει εάν θέλει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλλον με παρεξήγησε ο συνάδελφος. Και ίσως δεν κατάλαβα και πολύ καλά ούτε τι είπε ο Επίτροπος, ούτε τι είναι γραμμένο στην έκθεση. Γιατί εγώ αναφέρθηκα στην αξιοπιστία και εσείς αναφέρεστε σε διορισμούς. Για μένα είναι σημαντικό το περιεχόμενο των στατιστικών. Πολύ πιο σημαντικό από το πόσες γυναίκες συνεδριάζουν σε ένα όργανο συλλογικό. Για μένα η αξιοπιστία, η καλή δουλειά έχει προτεραιότητα. Και είπα πως θα ήταν ενδιαφέρον και σημαντικό να καλέσουμε σε ακρόαση τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, γιατί ήθελα να κάνω ερωτήσεις και μεθοδολογικού χαρακτήρα για το πώς γίνεται η συλλογή των δεδομένων. Μία πρόταση για συνεργασία ήταν και ελπίζω να το αντελήφθη σωστά όπως το εννοώ και ο Επίτροπος. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, σας αντελήφθημεν. Ο κύριος Μπάνκι έχει στήσει το λόγο τελευταίος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιόπιστες στατιστικές χρειάζονται τόσο οι αρμόδιοι για τη λήψη των αποφάσεων όσο και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ετών οφείλονται κυρίως σε φαλκίδευση δεδομένων σχετικών με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών οδήγησαν σε σημαντικά προβλήματα ο πρώην ε, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ακολουθώντας τα βήματα του Τσόρτσιλ ε, ε, χρησιμοποίησε τις στατιστικές που τον εξυπηρετούσαν καλύτερα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των στατιστικών και για να αναφερθώ σε έναν διακεκριμένο ε, και βραβευμένο με το βραβείο Νόμπελ στο Χαστή, ε, οι ωραίες στατιστικές είναι σαν τις πλάτες των γυναικών. Τις κοιτάμε για λίγη ώρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες. Ο Επίτροπος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις απόψεις που εκφράστηκαν στη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Πράγματι, η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στα πρόγραμμά μας εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά κάπου στην πορεία οι αρχικοί στόχοι χάθηκαν εν μέσω συζητήσεων. Και είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι το κείμενο το οποίο έχουμε αναχείρα σήμερα χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και αυτό άλλωστε αναγνωρίστηκε και από τον εισηγητή. Τα κράτη-μέλη είναι και αυτά διχασμένα και το Συμβούλιο δεν μπορεί να υποστηρίξει το κείμενο. Η ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται από τις χώρες τις οποίες οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίε είναι ήδη ε, επαγγελματικά ανεξάρτητες ε, και ε, χαίρονται ιδιαίτερα για τα εθνικά στατιστικά του συστήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό το οποίο επιθυμούμε με αυτή την πρόταση είναι να αποκατασταθεί η φιλοδοξία του στο αρχικό επίπεδο το οποίο είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τουλάχιστον κάτι το οποίο να πλησιάζει σε αυτούς τους στόχους και αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε η κυρία Γκάλ ε, για το Γενικό Διευθυντή της Eurostat, τον οποίο θα έπρεπε να ακούσουμε και εδώ και να σας πω ότι εμείς ε, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την ιδέα αυτή στα πλαίσια του διαφθορωτικού διαλόγου και επίσης να πω ότι μας ανησυχεί ιδιαίτερα και η ανεξαρτησία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και θέλουμε πραγματικά η οδηγία να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Οι δυνατότητες συντονισμού τους είναι ζωτική σημασία για τα αξιόπιστα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία και φυσικά ε, το όλο θέμα της αξιοπιστίας είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ ότι έχουμε κοινού στόχου. Αυτό λοιπόν που απαιτείται πλέον είναι να επεξεργαστούμε το θέμα λίγο περαιτέρω και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία πραγματικά θα διασφαλίσει ότι θα έχουμε υψηλή ποιότητα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία. Και εμεί από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε ένα τελικό συμβιβασμό και πραγματικά θεωρώ, πιστεύω ακράδαντα ότι το ίδιο θα κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή λύση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ τώρα τον εισηγητή να λάβει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, δικαίως είπατε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Και παρόλα αυτά, όπως είπατε, οι στόχοι μα είναι κοντά ε, με τους δε. Υπήρξε συμφωνία με τον άλλο συνομοθέτη από την 1η Ιουλίου με το Συμβούλιο, σχεδόν έξι μήνες πριν. Και ο ρόλος σας είναι να είστε και διαμεσολαβητές μεταξύ των συνομοθετών. Γιατί καθυστερείτε λοιπόν. Αύριο ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει μια στεναρή χειρονομία με την ψηφοφορία του που ελπίζω η Κομισιόν να τη λάβει σοβαρά υπόψη της. Γιατί η διαπραγμάτευση ελπίζω ότι θα συνεχιστεί και θα καταλήξει πολύ σύντομα. Ευχαριστώ τον Σίγητα. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση της εκθέσεως ψηφοφορία αύριο στις 12 το μεσημέρι και περνώ στο επόμενο θέμα της μέσης διάταξης έκθεση της κυρίας Στάινρουκ πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία Παρακαλώ τον να λάβει το λόγο.